Good morning, colleagues, and thank you to the... Καλημέρα συνάδελφοι. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που ήρθανε. καιρό. Μάλλον υπάρχουν κάποια προβληματάκια ε, με την απεργία στα μέσα συγκοινωνιών. Σας ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει, όσους ήρθατε. Και η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδικτύο. Οπότε να σας πω κύριε Σορέντερ ότι μας ακούνε από το διαδίκτυο τουλάχιστον. Ευχαριστώ παντού συναδέλφου που κατάφεραν να έρθουν. Οπότε ξεκινάμε με το πρώτο σημείο, το 15. Καλωσορίζω τον κύριο Ντέτλεφ Σρέντερ που έχει την πρώτη φορά εδώ ως νέος εκτελεστικός διευθυντής ε, του ΣΕΠΟΛ. Καλώς ήρθατε. Αναλάβετε τα καθήκοντά σας ε, στις 16 Φεβρουαρίου. Πριν ήσασταν υποδιευθυντής ε, και διευθυντής επιχειρήσεων επί σειρά ετών. Σήμερα λοιπόν θα μας ε, παρουσιάσετε τι έχει επιτύχει σε το 2017, το πρόγραμμα για το 2018 και τους ε, στρατηγικούς στόχους για το προσεχές μέλλον. Οπότε, έχετε τον λόγο για 10 λεπτά, έχετε την παρουσίασή σας και κατόπιν αν θέλουν και οι συνάδελφοι να κάνουν ερωτήσεις ε, μπορούν Καλώς ήρθατε λοιπόν και ακούμε την παρουσίασή σας. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την υποδοχή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι προνόμιο μου το ότι τα κράτη-μέλη μου έκαναν την τιμή να με ορίσουν εκτελεστικό διευθυντή της ε, ΣΕΠΟΛ και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας συναντήσω τόσο σύντομα και να σας παρουσιάσω κάποια αποτελέσματα από το 2017 και το τι αναμένουμε τα επόμενα χρόνια. Κάποιες παρατηρήσεις ε, και για εμένα. Επί 30 χρόνια ήμουν ε, αστυνομικός στην Γερμανία, επικεφαλής εγκληματολογικών τμήματων και περιφερειών τη αστυνομίας. Εδώ και 12 χρόνια βρίσκομαι στην υπηρεσία αυτή, την ΣΕΠΟΛ και χαίρομαι που θα έχουν ευκαιρία να ηγηθώ της υπηρεσίας τα επόμενα χρόνια. Να σας παρουσιάσω τώρα κάποιες βασικέ πτυχές για την στρατηγική μας, το πόσο βλέπουμε αυτούς, τι θέλουμε να προσφέρουμε στην ευρωπαϊκή κοινότητα να σας δώσω κάποια αποτελέσματα από τις δραστηριότητές μας το 2017 και μετά την πρόβλεψη για τα επόμενα έτη. Επόμενη διαφάνεια. Κάποιες βασικές πτυχές για τον ρόλο μας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε μια υπηρεσία πρώτης γραμμής, δηλαδή αν υπάρχουν κάποιες απειλές για την ευρωπαϊκή κοινότητα τότε πρέπει σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες δικαιοσύνης και εσωτερικών να προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη απάντηση για αυτές τις ε, απειλές. Γι' αυτό προσπαθούμε, έχουμε ένα εξαιρετικό εργαλείο για να μεταφράσουμε τις ε, πολιτικές δικαιοσύνης και εσωτερικών σε συγκεκριμένες δράσεις μέσω της εκπαίδευσης ε, και βεβαίως ο νόμος ε, που μόνος του μπορεί να είναι εξαιρετική ε, νομοθεσία αλλά θα πρέπει ακριβώς ε, να μπορέσουν στη δική μας περίπτωση να αντιληφθούν οι ιδιοκτικές αρχές το τι ακριβώς σημαίνει, με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν και με ποιον θα πρέπει να συνεργαστούν. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είμαστε το μέσο ακριβώς το οποίο θα βοηθήσει στην μεταφορά ε, των νομοθετημάτων αυτών στην πράξη μέσω της εκπαίδευσης ε, των αστυνομικών δυνάμεων. Υποστηρίζουμε λοιπόν ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω πολυεπίπεδων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να δώσουμε πολλαπλές ε, απαντήσεις Προσπαθούμε δηλαδή πρώτα απ' όλα να αναλύσουμε το πρόβλημα και μετά να σκεφτούμε είναι, ε, ποια είναι η καλύτερη απάντηση στον τομέα τη εκπαίδευση. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι πάντα η εκπαίδευση είναι η απάντηση. Εστιάζουμε στου βασικούς τομείς όπως η αντιτρομοκρατία, μετανάστευση, κύβερνο έγκλημα και σοβαρό εργανομένο έγκλημα. Και αυτό γίνεται πάντα σε πολύ στενή συνεργασία με όλε τι άλλε υπηρεσίε που λειτουργούν στον τομέα αυτό. Επίση προσπαθούμε να βρούμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τις διάφορες επιλογές ε, που έχουμε. Θα σας εξηγήσω μετά και το τι κάνουμε στον τομέα της ηλεκτρονικής διδασκαλίας που είναι ένα πάρα πολύ ε, φτηνό αλλά και γρήγορο και ευέλικτο εργαλείο. Προσπαθούμε λοιπόν να τα συνδυάσουμε αυτά με τρόπο αποτελεσματικό στο πλαίσιο του προπολογισμού μας. Εστιάζουμε εδώ και κάποια χρόνια στις ανάγκες ε, των επιχειρησιακών ε, κλάδων της αστυνομίας. Να ε, περάσουμε δηλαδή ακριβώς ε, στις ε, προτεραιότητες e ΕΜΠΕΚ και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο γύρω από αυτούς επόμενη διαφάνεια. Προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο ευέλικτοι απέναντι στι νέε απειλέ. Μπορώ να σα πω ότι τα τελευταία χρόνια, το έχετε συζητήσει σίγουρα, ε, οτιδήποτε αφορά την παράνομη μετανάστευση, την τρομοκρατία τα τελευταία χρόνια, όταν εμφανίστηκαν αυτά τα ζητήματα, αυτομάτως ε, αλλάξαμε και το πρόγραμμά μας για να στηρίξουμε τις επιχειρησιακές κοινότητες στην Ευρώπη όσον αφορά την εκπαίδευση την κατάρτιση, πώς θα αξιολογούμε τις ε, τρομοκρατικές απειλές, ε, τους ε, ξένους τρομοκράτες, μαχητές κτλ. Και ακριβώς να στηρίξουμε τις σχετικές κοινότητες της αστυνομίας. Επίσης, αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Ένωσης και την σχέση μεταξύ τους. Πώς το κάνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα είμαστε σε επαφή με τις περισσότερες χώρες ε, της γειτονία με όλες τις βαλκανικές χώρες, ε, ιδιαίτερως των Δυτικών Βαλκανίων. Συνεργαζόμαστε επίσης με χώρες στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική και προσπαθούμε εκεί πέρα να συνδυάσουμε τις διάφορες ανάγκες, να συνεργαζόμαστε με τις χώρες αυτές και επίσης ε, φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε, να συνεργάζονται και οι εταίροι μας εντός της Ένωσης με τους ομολόγους τους εκτός της Ένωσης ε, για πρώτη φορά. Αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα για να υπάρχει μια καλύτερη αντίληψη του ότι πρόκειται για ένα οριζόντιο στοιχείο που διατρέχει όλες μας τις δραστηριότητες και εκτός της Ένωσης αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο κράτος δικαίου σε χώρες όπως η Ορδανία, ο Λίβανος, η Τινησία πάντα τονίζουμε την δική μας ε, την πτυχή και αντίληψη του κράτους δικαίου. Επόμενη διαφάνεια. Ε, θεωρούμε επίσης ότι ο ρόλος μας ε, είναι να συνεισφέρουμε σε μια κοινή κουλτούρα επιβολής ε, του νόμου. Τι σημαίνει αυτό. Καθώς έχω μεγάλη εμπειρία στην διεθνή συνεργασία γνωρίζω πως αυτά τα πράγματα λειτουργούν μόνο αν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων εταίρων. Αν μιλάμε για ευαίσθητε έρευνε, π.χ. στο οργανωμένο έγκλημα ή στην τρομοκρατία, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη για να μοιράζονται οι υπηρεσίες πληροφορία. Και για να γίνει αυτό, είμαστε κι εμείς ένα εξαιρετικό εργαλείο, γιατί φέρνουμε τα άτομα σε επαφή όταν στέλνουμε, παραδείγματο χάρη, αστυνομικού από τη μία χώρα στην άλλη, βλέπουν με τα μάτια τους το πώς έχει η κατάσταση σε άλλους οργανισμούς, τι είναι δυνατόν, τι δεν είναι δυνατόν, ποιες είναι οι αδυναμίες και τα ισχυρά σημεία και έχουμε έτσι μια σωστή βάση ε, για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Επίση, κοινέ αξίε, όταν μιλάμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα, αυτά μπορούν να τα υποστηρίξουν οι εκπαιδευτικέ μα δραστηριότητε. Όπω ανέφερα και πριν, ε, συνεργαζόμαστε στενά με τους άλλους εταίρους μας ε, στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών ε, και από τη φάση του σχεδιασμού και οπωσδήποτε στην εφαρμογή. Να σας κάποια παραδείγματα. Στο 60% των δραστηριοτήτων μας ε, η Europol έχει άμεση εμπλοκή, συνεισφέρει όχι μόνο στις δραστηριότητες αλλά ήδη από την φάση του σχεδιασμού και της εφαρμογής και της συνέχειας προσπαθούμε να συνεργαστούμε. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες υπηρεσίες όπως η Frontex, η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κτλ. Επίσης θα ήθελα να τονίσω πως έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με την Κομισιόν, ειδικά την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών, γιατί παίζουν και αυτοί πολύ σημαντικό ρόλο και είμαι ευγνώμων για τα όσα έχουμε επιτύχει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού για το μέλλον προετοιμαζόμαστε για την αλλαγή νοοτροπίας ε, στον τομέα της εκπαίδευσης. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες, γιατί αλλάζει η κοινωνία, αλλά και ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Τώρα, ε, σήμερα εσείς ε, και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν πλέον τόσο πολλές πληροφορίες διαθέσιμες στο διαδίκτυο και η αντίληψη του τι εστί ε, γνώση και μάθηση αλλάζει. Εμείς λοιπόν ως οργανισμός έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση όσον αφορά την ηλεκτρονική μάθηση και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ πέρα βλέπετε τους συμμετέχοντες ε, στον τομέα της επιβολής ε, του νόμου στις δραστηριότητες μας. Το 2010 είχαμε 2.000 συμμετέχοντες ε, και βλέπετε τι πετύχαμε πέρσι. Είχαμε σχεδόν 24.000 συμμετέχοντες στις δραστηριότητες μας. Χαιρόμαστε με αυτήν την αύξηση η οποία κατέστη δυνατή ε, χάρη στη μεγάλη χρήση ηλεκτρονικής εκπαίδευσης γιατί είναι ένα πολύ ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο ε, βεβαίω δεν μπορεί να αντικαταστήσει την φυσική παρουσία οπωσδήποτε, αλλά τα νούμερα αυτά σας δίνουν μια εικόνα του πώς ε, έχει αυξηθεί η δραστηριότητά μας, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερα στο μέλλον για να έρθουμε σε επαφή και με άλλες ε, ομάδες. Λοιπόν, επόμενη διαφάνεια. Εδώ πέρα βλέπετε παράλληλα την εξέλιξη του προϋπολογισμού της υπηρεσίας μας. Ε, βλέπετε ότι έχουμε λίγο πολύ τον ίδιο προϋπολογισμό, μία μικρή αύξηση το 2017, φέτος έχουμε μία μικρή μείωση, βλέπετε όμως ότι παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει να έρθουμε σε επαφή με πολύ περισσότερους. Επόμενη διαφάνεια, να σας δώσω κάποια νούμερα για το τι κάνουμε συγκεκριμένα στους συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητες. Στην αντιδρομοκρατία έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από χίλιους, σχεδόν 1100 αστυνομικούς για θέματα μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης, επίσης γύρω στα 1000 άτομα, 909. Ε, Κυβερνοέγκλημα, κυβερνοασφάλεια, θα επανέλθω. Πέρσι εκπαιδεύσαμε 4.450 αστυνομικούς ε, και εδώ πέρα αυξάνεται η ζήτηση σε άλλους τομεί, ε, σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Εκπαιδεύσαμε πέρσι γύρω στα 5.000 άτομα και δείχνουμε εδώ πέρα πως η ΣΕΠΟΛ ε, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην ζήτηση που υπάρχει για εκπαίδευση στους ε, επιχειρησιακούς τομείς με τον καλύτερο τρόπο και δεν είναι θέμα μόνο ποσοτήτων, μπορώ να σας πω ότι μετράμε πάντα και αξιολογούμε όλες τις δραστηριότητες αν ανταποκρίνονται ανάγκες και αν οι πελάτες μας είναι ικανοποιημένοι. Και πάντα έχουμε ένα ποσοστό ικανοποίησης πάνω από το 90%, κατά κανόνα 93-94% των συμμετεχόντων. Συνεργαζόμαστε, όπως σας είπα, και με χώρες της ε, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Και μάλιστα πέρυσι ε, έχουμε ένα σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή αυτή για την αντιτρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη και αντιληφθήκαμε και εμείς την ανάγκη να ενδύνουμε τις προσπάθειές μας και να συνεργαστούμε πιο στενά με τις χώρες Μέση Ανατολής και Βόρειας Αφρικής και να τις βοηθήσουμε, να τις ενδράμουμε για να αντιμετωπίσουν τα πολλά προβλήματα που έχουν. Είχαμε αγαστή συνεργασία με τέσσερις χώρες, Τουρκία, Λίβανο, Ιορδανία και την Ισία και βλέπετε πόσους ε, υπαλλήλους εκπαιδεύσαμε. Και μάλιστα οι χώρες αυτές έχουν εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέρον για στενή συνεργασία με τις ε, ευρωπαϊκές κοινότητες ε, ε, ομάδες επιβολής του νόμου. Και μάλιστα στην περίπτωση της Τουρκίας, βέβαια η καιρή στη συνεργασία είναι κάπως πιο απαιτητική και πιο δύσκολη, αλλά έχουμε συνεννόηση και κοινή αντίληψη των δραστηριοτήτων που πρέπει και των επιχειρήσεων που πρέπει να εφαρμόσουμε. Σε ό,τι αφορά το μέλλον 2018-2020. Καταρχήν, εγώ ως εκτελεστικός διευθυντής προσβλέπω στην ε, πλήρη υλοποίηση της νέας ε, εντολής που έχουμε αναλάβει από το 2016 και εκτιμούμε ιδιαίτερο στη διευρυμένη εντολή που δώσατε στην Αστυνομική Ακαδημία και θέλουμε να την αξιοποιήσουμε και να την εφαρμόσουμε στο έπακρο. Βέβαια, πολλές δράσεις ακόμη θα πρέπει να επιτελεστούν. Καταρχήν, ε, θέλουμε ε, να προσφέρουμε προσαρμοσμένες τις ειδικέ ανάγκες ε, των ε, αστυνομικών αρχών δραστηριότητες και επίσης να συμβάλλουμε σε καλύτερο συντονισμό. Γιατί έχουμε τελωνιακές αρχές, διοκτικές αρχές, αστυνομικές αρχές, και θα προσαρμόσουμε την προσφορά μα στι ανάγκε των κρατών μελών. Επίση, θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα για καλύτερο συντονισμό τη εκπαίδευση ε, των ε, αρχών επιβολή του νόμου στην Ευρώπη. Θέλουμε στενότερη συνεργασία σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και κάποιοι εξωτερικοί οργανισμοί έχουν τις τη δική του εντολή σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και σεβόμαστε απόλυτα αυτέ τις εντολές, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το συντονισμό και να το καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό στο μέλλον, ώστε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και να έχουμε το βέλτιστο συντονισμό αξιοποιώντας τις συνέργειε που υπάρχουν σε ορισμένου τομεί. Και μάλιστα στο, τον περασμένο χρόνο το συζητήσαμε με τις ε, με τους αρμόδιους οργανισμούς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εμπλέκεται ενεργά σε αυτό το μηχανισμό βελτίωσης του συντονισμού. Και εδώ έχουμε κάποια απτά παραδείγματα. Καταρχήν ε, θα, θα διευρύνουμε το πρόγραμμα των ανταλλαγών στη συνεργασία με τη Frontex και θα έχουμε κάποιες ε, βελτιώσεις στην διοικητική διαχείριση των προγραμμάτων με κάποιες ε, ε, Συγχωνεύσει και αξιοποίηση του δυναμικού και σε άλλους τομείς. Τώρα, στο μέλλον θα θέλαμε καλύτερη ανάπτυξη των ε, κέντρων γνώσης της ΣΕΠΟΛ. Ξεκινήσαμε με δύο κέντρα γνώσης ε, σε άλλους τομείς τους, αποκαλούμε κέντρα αριστείας. Εμείς είμαστε πιο μετριόφρονες, τους αποκαλούμε κέντρα γνώσης. Προσβλέπουμε βέβαια να γίνουμε κέντρα αριστείας. Και μάλιστα τώρα επικεντρωνόμαστε σε δύο θέματα, στην αντιτρομοκρατία και στήριξη ε, των αποστολών ε, της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Θέλουμε μια βιώσιμη ε, ανάπτυξη και συνεργασία και μάλιστα δεν έχουμε μόνο ετή συνεργασία αλλά πολυετή. Και μάλιστα προσπαθούμε με εφόρο τρόπο να επιτρέψουμε στους εταίρους μας να αναλάβουν την ευθύνη και να κάνουν κτήμα τους αυτές τις δράσεις. Και έχουμε το κέντρο τρομοκρατίας της ε, Europol και σε ό,τι αφορά τις αποστολές ε, CSDP ε, προσπαθούμε να εμπλέξουμε και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στα θέματα αυτά. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα συνεργασίας. Και περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. το κυβερνοέγκλημα και τα συνεφή εγκλήματα του κυβερνοχώρου. Ε, δίνουμε ιδιαίτερα προσοχή σε αυτά τα θέματα γιατί υπάρχει μεγάλο αίτημα των κρατών μέλων ε, για βοήθεια σε θέματα εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και συναφή εγκλήματα. Και φυσικά σίγουρα τα κυβερνοεγκλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει ανάγκη διασυνοριακής ε, συνεργασίας και έχουμε κάποιες διεθνείς ε, δραστηριότητες εκπαίδευσης. Και μάλιστα κάθε χρόνο θέλουμε ανανέωση της εκπαίδευσης, γιατί είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις ε, στο κυβερνοέγκλημα που και η εκπαίδευση θα πρέπει να ακολουθεί. Και μάλιστα λόγω του μεγέθους των επενδύσεων, τα κράτη-μέλη από μόνα τους δεν μπορούν να, να παρακολουθήσουν το ρυθμό ανάπτυξης του κυβερνοέγκληματος και να έχουν καλά καταρτισμένους ε, εμπειρογνώμονες. Και σίγουρα όταν υπάρχουν τέτοιοι οι δήμονες, ε, τους προσελκύει ο ιδιωτικός τομέας ε, που έχει καλύτερες αμοιβέ. Γι' αυτό και πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη σε τέτοιου είδους θέματα εκπαίδευσης για το κυβερνοέγκλημα σε συνεργασία με το αντίστοιχο κέντρο της Ευρωπόλ. Ε, επίσης, θέλουμε μεγαλύτερη έμφαση της εξωτερικής διάσταση της εσωτερική ασφάλειας. Στηρίζουμε καλύτερα τις αποστολές, ε, κοινές αποστολές ε, ε, ασφάλειας και άμυνας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ικανότητες και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ένα άλλο σχέδιο στη Μένα, περιοχή Μένα, καλύπτοντας και την Αλγερία και το Μαρόκο πέραν των υπόλοιπων χωρών Μέση Ανατολής και Βορειοαφρικής και έχουμε και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα στα Δυτικά Βαλκάνια. Είμαστε βέβαιοι ότι ε, έχουμε σχετικά ισχνές ε, δομές διοικητικές και δημοσιονομικές. Έχουμε ένα 95% ποσοστό ε, δέσμευσης και μια αποκεντρωμένη ανάπτυξη προκειμένου να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και να αξιοποιήσουμε τις δομές των κρατών μελών και μάλιστα 70% των ε, σεμιναρίων μας γίνονται σε πανεπιστήμια, σε ακαδημίες, σε κολέγια, στα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη διενεργούν αυτές τις δραστηριότητες εκ μέρους μας, ε, δίνοντας, προσδίδοντας μία ευρωπαϊκή διάσταση. Και έτσι στηρίζουμε και τη συμμετοχή άλλων εταίρων από άλλα κράτη-μέλη. Επίσης, πρωτοστατούμε στην παροχή προγραμμάτων ανταλλαγής υπαλλήλων ε, των αστυνομικών και διεκτικών αρχών και φυσικά αξιοποιούμε καλύτερα την ηλεκτρονική μάθηση αξιοποιώντας ε, τα προγράμματα εκπαίδευσής μας και τις τεχνολογικές δυνατότητες. Και προσφέρουμε και σε άλλους εταίρους τεχνικές, τεχνολογικές πλατφόρμες που μπορούν να τις αξιοποιήσουν για τις δικές τους δραστηριότητες. Όπως είπα και προηγουμένως, σε ό,τι αφορά κάποια στοιχεία της ε, εκπαίδευσης των αστυνομικών και διεκτικών αρχών, ε, τα κράτη-μέλη μερικές φορές έχουν δυσκολίες να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στους υπαλλήλους τους. Ιδιαίτερα οι μικρότερες χώρες ε, αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να υποστηρίζονται από τις ευρωπαϊκές δομές. Βέβαια θα πρέπει να μεριμνούμε ώστε να, να ενισχύουμε τους πιο αδύναμους κρίκους της αλυσίδας ό,τι αφορά τις απειλές της εσωτερικής ασφάλειας. Γι' αυτό και θα πρέπει να δίνουμε τις προσπάθειές μας και να στηρίξουμε τους εταίρους που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν κατάρτιση υψηλού επίπεδου. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση από τα κράτη-μέλη και τις διάφορες κοινότητες και μάλιστα και τα τελωνία, ε, οι υπάλληλοι τελωνίων ζητούν υποστήριξη από τις ΣΕΠΟΛ στο μέλλον. Γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχύσουμε και εδώ τις προσπάθειές μας. Αυτά από πλευράς ΣΕΠΟΛ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και πολύ ευχαριστώ να απαντήσω στις απορίες σας και να δώσω περισσότερες πληροφορίες για την Ακαδημία μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σρόντερ. Νομίζω ότι ιδίως με ε, την υπηρεσία σας είναι πολύ σημαντικό να φωτίζονται αυτά τα ζητήματα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνονται επισκέψεις. Ε, έχουμε και μια αποστολή τον ε, Απρίλιο που θα σας επισκεφθεί ε, και νομίζω θα είναι πολύ θετικό προκειμένου να αποκτήσουν τα μέλη της Επιτροπής μας μια καλύτερη εικόνα για τα επιτεύγματά σας στην υλοποίηση της στρατηγικής σας. Θέλει κάποιο μέλος της Επιτροπής να πάρει τον, το λόγο, κύριε Σιππελ. Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση, κύριε Στρέντερ. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Τα τελευταία χρόνια κάναμε πολλά βήματα για να εναρμονίσουμε κατά κάποιο τρόπο το έργο, αλλά κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών ε, οδηγιών αλλά και της εθνικής νομοσίας υπάρχουν πολύ, πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πώς χειρίζεστε, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα στη ΣΕΠΟΛ ή μήπως επικεντρώνεστε μόνο στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αν και νομίζω ότι αναγκαστικά σας επηρεάζει. Επίσης, το έργο σας αυξάνει την κατανόηση των διαφόρων συστημάτων, ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών και δικαστικών αρχών. Επίσης, για τις κοινέ ε, ε, ομάδες διερεύνησης, ε, πολλοί αστυνομικοί μου έχουν πει ότι έχουν αποκομίσει πολύ θετικές εμπειρίες από αυτό. Το ερώτημα μου είναι, το έργο της ΣΕΠΟΛ βοηθά, ενθαρρύνει τους αξιωματούχους ώστε να δραστηριοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν, ε, υπάρχουν αξιωματικοί πολιτικοί οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδου ομάδε χωρί να έχουν παρακολουθήσει ε, εκπαιδευτικού κύκλου τη ΕΠΟΛ ή πρέπει πρώτα να έχει κανεί παρακολουθήσει κατάρτιση τη ΕΠΟΛ και στη συνέχεια να συμμετέχει σε τέτοιου είδου ομάδε. Για την συνεργασία σα με χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρατε ότι επικεντρώνεστε στο κράτο δικαίου. Θυμάμαι ότι σε μία από τις παλαιότερες συναντήσεις μας κάποιος μας είχε πει ναι εντάξει το κράτος δικαίου είναι καλό αλλά ακόμη και δικτάτορες μπορεί να εφαρμόζουν το κράτος δικαίου εφαρμόζοντας το δίκαιο των χωρών τους. Ποιες είναι λοιπόν οι προκλήσεις ε, όταν μιλούμε για την εφαρμογή του κράτους δικαίου και ιδίως υπό τη σκοπιά της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και μια τελευταία ερώτηση. Μιλώντας για τις βασικές προτεραιότητές σας, ε, αποδεικνύεται ότι ε, υπάρχει ιδιαίτερη επικέντρωση από τα κράτη-μέλη στο κυβερνοέγκλημα και την κυβερνοασφάλεια. Υπάρχουν ιδιαίτερες πτυχές αυτού του τομέα στις οποίες επικεντρώνεστε και μια πραγματικά τελευταία ερώτηση. Μιλώντας για την ενισχυμένη ε, συμμετοχή στις εργασίες της ΕΠΟΛ, αυτή η αύξηση που υπάρχει προέρχεται από όλα τα κράτη-μέλη ή υπάρχει κάποια ανισορροπία ω προ την αύξηση αυτής τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Σόφι Ιντβελ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη γιατί έχασα το πρώτο κομμάτι της παρουσίασής σας. Το ερώτημα μου ε, αφορά κάτι που ενδεχομένως έχετε ήδη ε, απαντήσει, αλλά ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε κάποιες πληροφορίες για μια άλλη διάσταση της αστυνομικής κατάρτισης ε, που είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αφενός γνωρίζουμε ότι ε, και στις αστυνομικές αρχές υπάρχει ξενοφοβία, σεξισμός, ομοφοβία. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές είναι ε, εκείνες οι αρχές στις οποίες πρέπει να καταγγέλλονται εγκλήματα μίσους κτλ. Έχω αποστείλει στην υπηρεσία σας πολλές επιστολές ε, ρωτώντας για αυτά τα θέματα γιατί ε, ξέρω ότι όταν μεταφερθήκατε στη Βουδαπέστη υπήρχε αστυνομική αρχή εκεί στη Βουδαπέστη η οποία ε, έλεγε στις γυναίκες να μην φοράνε μήνυ όταν πηγαίνουν στα μπαρ γιατί αλλιώς ε, θα, είναι εκείνες που θα ευθύνονται για το βιασμό τους σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ελπίζω να έχουν βελτιωθεί λοιπόν τα πράγματα. Τι προγράμματα έχετε, όχι γενικά, τι κάνετε στην πράξη συγκεκριμένα ε, όσον αφορά την εκπαίδευση των αστυνομικών στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ, Σοφή. Να προσθέσω και εγώ κάτι για την επιβολή του νόμου και τη σχετική κατάρτιση. Τις προδιαγραφές που εφαρμόζονται στις αστυνομικές πρακτικές, στη διαφθορά, με την ευρύτερη έννοια. Η δωροδοκία, για παράδειγμα, τέτοιου είδου θέματα. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς λοιπόν είστε στην υπηρεσία αυτή εδώ και πολλά χρόνια. Ποια είναι η αίσθησή σας, πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι διαφορές, ποιες είναι οι πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Συνδέεται και με το ερώτημα της Όφης, γιατί αν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν βελτιώνεται, τότε αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως εφαλτήριο για ε, διακρίσεις. Ακριβώς γιατί μειώνονται τα οι προδιαγραφές. Ποια είναι η αίσθησή σας. Δουλεύετε πολλά χρόνια στην υπηρεσία. Τα πράγματα βελτιώνονται ή μήπως ε, το πολιτικό κλίμα που επικρατεί σε κάποιες χώρες τουλάχιστον επιδεινώνει τα πράγματα. Υπάρχουν ε, καλές πρακτικές χωρίς να θέλω να αποκαταλάβω την απάντησή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Πρώτον, πώς προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε και με την Eurojust και με το δικαστικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, σκοπός μας είναι πάντοτε να αξιοποιούμε βεβαίως τα ενωσιακά εργαλεία, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και εθνικά και διεθνή ε, εργαλεία και μηχανισμοί. Χρησιμοποιούμε λοιπόν να ε, εφαρμόζουμε μια οριζόντια προσέγγιση στη συνεργασία αστυνομικών και δικαστικών αρχών και γι' αυτό μας ενδιαφέρει πολύ η συνεργασία και με τους ε, φορείς που δρούν επιτόπου. Πρέπει να σας πω όμως ότι αυτό που με εντυπωσιάζει πολλές φορές, καθώς προέρχομαι και από μια εθνική αρχή όπου υπήρχε στόχος να υπάρχει συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών, εισαγγελείς, δικαστές, τότε ε, όταν εγώ τουλάχιστον ήμουν ήταν πολύ δύσκολο να υπάρχει κοινή συνεδρίαση. Υπήρχαν όμως δίκτυα όπου συγκεντρώνονταν ε, άνθρωποι και από τις δύο ε, πτυχές ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για το ποιες, είναι οι προκλήσεις και να συζητούνται ε, λύσεις των προβλημάτων. Για τις κοινέ ε, ομάδες ερευνών υπάρχουν προπαρασκευαστικές ε, ε, εκπαιδευτικές μονάδες, κύκλοι για αστυνομικούς και δικαστικούς υπαλλήλους Υπάρχει, έχουν στεφτεί με επιτυχία αυτές οι διαδικασίες υπάρχει μεγάλη αύξηση της συμμετοχής και αστυνομικών και δικαστών προκειμένου να προετοιμάζονται και οι δύο πλευρές για αυτά τα τζιτς και βλέπουμε ότι ε, έχουν, ε, υπάρχουν θετικά ε, ωφέλη και στην εφαρμογή αυτών των ερευνών, στην υλοποίηση και στη δραστηριοποίησή τους και θα σας δώσω και υπάρχουν και παραδείγματα όπου δημιουργήθηκαν τέτοιες ομάδες και στα Δυτικά Βαλκάνια. Υπήρχαν λοιπόν αξιωματούχοι και από την Ευρώπη και από τα Δυτικά Βαλκάνια κατά την, το σχεδιασμό αυτών των ζήτων. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε είναι κάποιες φορές να υπάρχει ε, ε, ανάγκη να δημιουργηθεί μια τζιτ και να στελεχωθεί με ε, ανθρώπους που δεν έχουν λάβει κατάρτιση από εμάς. Ε, Ιδίω όμως στα Βαλκάνια υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τη δημιουργία τέτοιων κοινών ομάδων και τη συνεργασία. Είναι λοιπόν ένα θετικό εργαλείο το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα στο μέλλον και εμείς υποστηρίζουμε στο μεγαλύτερο, στο, στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις εκπαιδεύσεις γύρω από αυτό. Είπατε πώς ενισχύουμε την εμπιστοσύνη και πώς μπορεί αυτό να γίνει από τη δική μας πλευρά με συγκεκριμένα μέτρα. Το να συγκεντρώνονται λοιπόν άτομα και στις εκπαιδεύσεις μας και στα online εργαλεία μας. Νομίζω το καλύτερο παράδειγμα είναι τα ε, προγράμματα ανταλλαγής. Είναι εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να μπορεί καθένας να ε, αποκτά μια μικρή απόσταση από το εθνικό του περιβάλλον ε, όταν έρχεται λοιπόν κάποιο, βλέπει ότι υπάρχουν και άλλε αστυνομικέ αρχέ οι οποίε δρούν διαφορετικά, όχι καλύτερα, όχι χειρότερα, έχουν όμω διαφορετικό νομικό πλαίσιο, διαφορετικέ συνθήκε εργασία, ακόμα και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται είναι διαφορετικό και αυτό βοηθά προκειμένου να αποκτά κανεί μια καλή αντίληψη για την συνεργασία. Και αυτός, αυτή η προσωπική διάσταση ε, του ότι έχουν επαγγελματίε δηλαδή τη δυνατότητα να μιλούν μεταξύ του. Ε, είναι πολύ θετική. Βλέπω ότι αυτό πολλές φορές δρά πολύ θετικά, γιατί μπορεί κανείς να μάθει και από τον συνάδελφο του από μια άλλη χώρα. Είναι, δηλαδή, υπάρχει λοιπόν τυπική διάσταση, αλλά υπάρχει και αυτή η μη τυπική διάσταση της προσωπικής, ας πούμε, επαφής, η οποία βοηθάει. Το άλλο στοιχείο που αναφέρατε, τι γίνεται ε, όσον αφορά τις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς και είναι πρόκληση αλλά την αντιμετωπίζουμε, την παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά αυτή την πρόκληση και είναι, ε, πρέπει να σας πω ότι στις δραστηριότητε μας στην Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική αποτελεί προτεραιότητά μας και από ό,τι θυμάμαι ε, Έχουμε προσκαλέσει και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων προκειμένου να κάνουν παρουσιάσεις στις εκπαιδεύσεις μας. Ε, και αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αξιωματούχοι αυτών των χωρών είναι τουλάχιστον ανοιχτοί στο να ακούσουν ποιες είναι οι δικές μας αντιλήψεις, ποια είναι η δική μας νοοτροπία και ε, πρέπει να ξέρετε ότι η κατάσταση στις διάφορες χώρες αυτές είναι και πολύ διαφορετική. Όταν μιλούμε για την τρομοκρατία, στο Λίβανο και στην Ιορδανία, για παράδειγμα, οι αξιωματούχοι, οι αστυνομικοί έχουν ε, πολύ διαφορετικό όγκο προκλήσεων και προβλημάτων να αντιμετωπίσουν. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει στο να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς την, ε, την άποψή μας για το ποια είναι η, η θέση μας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το, το κράτος δικαίου και πρέπει να είναι διάσταση των ε, ερευνών και των δραστηριοτήτων ε, είναι λοιπόν προτεραιότητά μας. Βεβαίως δεν ε, αντιλέγω ότι είναι πρόκληση για μα. Υπάρχουν διαφορετικές ε, κοινωνικές, ιστορικές συνθήκες, ιστορικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο στη δραστηριότητα αυτή. Για το κυβερνοέγκλημα, κυβερνοασφάλεια. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να έχουμε πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής μας ότι είναι ένα πολύ ευρύ θέμα ε, περιλαμβάνονται πάρα πολλά θέματα. Βεβαίω, οι μικρέ χώρε πρέπει να προστατεύονται ε, και να προετοιμάζονται καλύτερα ε, αλλά και ευρύτερα όπω οι πληροφορίες ανοιχτή ανοιχτής πηγής εκεί εκεί έχουμε διοργανώσει τρεις εκπαιδεύσεις Παρά το γεγονό ότι είχαμε αρχικά προγραμματίσει να κάνουμε μόνο μία, ακριβώ γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ε, γιατί είναι σημαντικό να, να, ε, μπορεί κανείς να αξιοποιήσει ε, ε πληροφορίες που είναι δημόσια ε, προσβάσιμες από το, το, το ίντερνετ. Προσπαθούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε μια διαρθρωμένη προσέγγιση και σε συνεργασία με την Ευρωπόλ προκειμένου να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι, ποιε είναι οι προκλήσει, τι πρέπει να επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια. Και ω ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό βεβαίω δρούμε πάντοτε συμπληρωματικά. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τι βασικέ δομέ που υπάρχουν και ε, εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Για την συμμετοχή από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τις ε, τις, ε, τις εκπαιδεύσεις μας και τα, τα, προγράμματα αντιληγής υπάρχει ε, ίση συμμετοχή και ζήτηση από τα κράτη-μέλη. Και ε, βλέπουμε μάλιστα ότι οι πόροι μας δεν επαρκούν για να καλύψουμε τη ζήτηση που υπάρχει και, στο, και στις πληροφορίες ε, ανοιχτής πηγής υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι μπορούμε εμείς να καλύψουμε. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά μέσα ε, βλέπουμε μεγάλη διακύμανση μεταξύ των κρατών μελών ε, ως προς την αξιοποίηση των υπηρεσιών μας. Κάποια κράτη-μέλη ε, πολύ ενεργά ε, ε, συμμετέχουν, κάποια λοιπόν αξιοποιούν αυτές τις υπηρεσίες, κάποια άλλα κράτη-μέλη, ακόμη και για τεχνικούς λόγους, ενδεχομένως γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τα, τους υπολογιστούς από τα γραφεία τους, δεν δραστηριοποιούνται τόσο πολύ, αλλά εργαζόμαστε και επί πρακτικών λύσεων. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ε, σκεφτόμαστε ενδεχομένως να, μπορέσουμε, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ε, συμμετρικό, το οποίο θα αντικατοπτρίζει τη δική μας δουλειά ε, απλά μέσω των, ε, των εθνικών ε, δικτύων. Επίσης, με τις διάφορες πτυχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων συμφωνώ απολύτως μαζί σας είναι πάρα πολύ σημαντικές για την εκπαίδευση και θα θυμάστε ότι πέρσι είχαμε και μια εκδήλωση σε αυτό το κτίριο Έχουμε ειδικέ δραστηριότητε για τα εγκλήματα μίσου, έχουμε σχετική εκπαίδευση, έχουμε εκπαίδευση των εκπαιδευτών για τα θεμελιώδη δικαιώματα, στο διαδίκτυο επίση. Και γνωρίζω ότι σα χρωστάω ακριβώ και το κομμάτι το online. Οπότε το παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά, όπως είχα επισημάνει όπως εμείς το βλέπουμε προσπαθούμε σε κάθε δραστηριότητα να δούμε το ποιο στοιχείο των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να τονίσουμε. Π.χ. όταν μιλάμε για σεξουαλική εκμετάλλευση στο διαδίκτυο είναι σαφές πως έχει ακριβώς μεγάλη σημασία το να μιλάμε για την προστασία των παιδιών ή για άλλες δραστηριότητες όπως η για αλλε δραστηριοτητε οπως στοιχείων στον δρόμο. Ξέρουμε πως δεν υπάρχει μια κοινή προδιαγραφή στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να δούμε τα καλά παραδείγματα και τα παρουσιάζουμε αλλά και εκεί ελπίζω με τον τρόπο που τα παρουσιάζουμε κάποιος από, εκτός της κοινότητας να σκεφτεί ότι αν ναι, αυτό στη χώρα το κάνουν διαφορετικά, ίσως είναι κάτι πιο καινούριο, πιο αποτελεσματικό, γιατί βέβαια το θέμα δεν είναι μόνο το τι κάνουμε ή το πώς ερευνούμε το έγκλημα, αλλά και το πόσο ανοιχτοί είμαστε απέναντι στις ε, διαφορετικές στοιχείες ε, των εγκληματών μίσους, πόσο ευαίσθητοι, προσπαθούμε να τα δούμε αυτά και όπως είπατε επίσης αυτή τη στιγμή ε, βλέπω πως υπάρχει κάποιος κίνδυνος, βλέπω κάποιες πολιτικές τάσεις που θα έρθουν αργότερα και στην επιβολή του νόμου, που σημαίνει ότι θα έχουμε χαμηλότερη προτεραιότητα σε αυτό το τομέα, κάτι το οποίο θέλω να αποφύγουμε. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ειδικά οι δραστηριότητες εκπαίδευσης ε, των εκπαιδευτών. Είχαμε κάνει πέρσι μία στην Αυστρία ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο γιατί ακριβώς ε, μπορούμε να έχουμε έτσι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιρροή. Αυτό το οποίο είπατε για τις διαφθορές, την διαφθορά με συγχωρείτε, για τις πρακτικές της αστυνομίας αυτό το οποίο κάνουμε υπάρχουν ε, βεβαίως ε, και σχετικές δραστηριότητες οποίες περιλαμβάνουμε την διαφθορά. Δεν έχουμε κάτι ειδικό για την διαφθορά. Ξέρω βεβαίως ότι αφορά πολλές κοινότητες ε, στην Ευρώπη. Εκεί πέρα θεωρώ ότι ο ρόλος μας είναι ότι πρέπει να πείθουμε μέσω των παραδειγμάτων του πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Και για μένα πάντα αυτό ξεκινάει στο επίπεδο των αξιών. Ποιος είναι ο ρόλος των αστυνομικών δυνάμεων σε κάθε χώρα. Είναι λοιπόν θέμα αξιών, κοινών αξιών και εκεί πέρα βλέπουμε τον ρόλο του ευρωπαϊκού επίπεδου, δηλαδή αυτό το οποίο, αυτό το οποίο αποφασίσαμε ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φτάνουν και στις ε, κοινότητες των αστυνομικών. Και μια τελευταία παρατήρηση πάντα εμείς ε, αναζητούμε την συνεργασία της Υπηρεσίας Θεμελιδών Δικαιωμάτων στην Βιέννη για να μοιράσουν και το υλικό τους ε, και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε καλύτερη επαφή και πρόσβαση στο εξαιρετικό υλικό τους. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Σρέντα, ευχαριστώ για την αναλυτική παρουσίασή σας. Είστε πολύ έμπειρος πράγματι και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον και σας ευχαριστώ που αναγνωρίζετε ότι θα υπάρχουν κάποια ζητήματα στο μέλλον αυτό το οποίο είπε η κυρία Ινετφέλντ. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ τους συναδέλφους που παρέμειναν ε, για την παρουσίασή σας η οποία βεβαίως μεταδόθηκε και στο διαδίκτυο. Δύσκολα τα ζητήματα νομίζω. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για τις ε, ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ και για την ε, παρουσίασή σας. Θα έχουμε και μία αποστολή της Επιτροπής μας στην Βουδαπέστη φέτος. Τώρα έχουμε τον πίνακα βαθμολογίας ε, και την έκθεση της κυρίας Κιγιώμη, η οποία θα έρθει στις 10 όμως. Έρχεται. Ευχαριστώ που έχουν έρθει οι σκιώδες εισηγητές και οι σόφοι. Έχουμε 10 λεπτά. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Και σόφοι, έχω να συζητήσω κάτι μαζί σας. Ε, ζητώ συγγνώμη για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, διάλειμμα λίγων λεπτών. Μέχρι να έρθει η εισηγήτρια για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Στέπερ. AUTHORWAVE Ευχαριστώ για την υπομονή σας αγαπητοί συνάδελφοι. Κατέφθασε η συγκεκριά μας, η κυρία Σελβί Γιώμ. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 των πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης. Όπως ξέρετε, δυνάμει το άρθρο 54, η Επιτροπή μας ε, είναι συνδεδεμένη επιτροπή και θα συμμετάσχει στην εκ, εκπόνηση της ε, έκθεσης Επιτροπής Γιούρι. Έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για τον πίνακα αποτελεσμάτων στην ποινική δικαιοσύνη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κοινέ ε, αρμοδιότητες ό,τι αφορά τι πτυχέ ε, του κράτου δικαίου. Η κυρία Γκυγιόμ θα μα ενημερώσει για τι τελευταίε εξελίξει και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Σε ευχαριστούμε Σιλβί που ήρθε Και το λέω ναι. Λόγω των δυσκολιών σήμερα. Παρακαλώ κυρία Γκυγιώμ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που περιλάβατε το σχέδιο εκθεσής μου στην ημερήσια διάταξη. Όπως γνωρίζετε, όπως μάλλον γνωρίζετε, πρόκειται για ένα πίνακα αποτελεσμάτων που από το 2013 δημοσιεύεται ετησίως και αφορά την αστική, εμπορική ε, και διοικητική δικαιοσύνη. Η ποινική δικαιοσύνη αποκλείεται. Θα επανέλθω στο σημείο αυτό αργότερα. Στόχος ε, του πίνακα αποτελεσμάτων είναι να βελτιώσει το ευρωπαϊκό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, δημιουργώντα ένα πρόσφορο έδαφος και ένα ευνοϊκό κλίμα για τις επιχειρήσεις, ε, τους καταναλωτές, ε, τους πολίτες γενικώ στα θέματα της δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά την ε, γνωμοδότηση της ΛΥΜΠΕ, εγώ επικεντρώθηκα στις αρμοδιότητες επιτροπής μας και κυρίως στην εξέταση του κράτους δικαίου. Επίσης, είναι σημαντικό στους μελλοντικούς πίνακες αποτελεσμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκύψει τα θέματα αυτά, προτείνοντας δείκτες για την αξιολόγηση του κράτους δικαίου. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εκπονήσει κάποιους δείκτες για το πώς τα κράτη-μέλη ε, διεκπεραιώνουν κάποιες παραβιάσεις που πλήττουν το κράτος δικαίου. Επίσης, ε, θα μπορούσαμε να λάβουμε κάποιο υπόψη κάποιες μορφές εγκληματικότητα που επηρεάζουν τον τρόπο απονομή τη δικαιοσύνης. Τρομοκρατία για παράδειγμα, αλλά όχι μόνο. Ας μην ξεχνούμε και τα θέματα νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητες. Επίσης το θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης ε, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του πίνακα αποτελεσμάτων. Και κάτι που μας είναι προσφυλές ε, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάγκη να υιοθετήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό μόνιμης ε, εποπτείας ε, της δημοκρατίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Και μάλιστα αυτό ήταν το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αποτυπώθηκε σε μια έκθεση πρωτοβουλία του 2016. Καλό θα ήταν λοιπόν να επαναλάβουμε την έκκλησή μας και την προτροπή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα μόνιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό. Βέβαια, επειδή είμαστε περιορισμένη στην έκθεση της γνωμοδότησης, δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε όλα. Πάντως, η ε, κυρία Γκέρτλαντ, που είναι η αρμόδια επί της ουσίας ε, στην έκθεση της Γιούρη, έχει περιλάβει στην έκθεση της πολλά σημαντικά σημεία. Εγώ στη γνωμοδότησή μου επικεντρώνομαι στο ζήτημα του κράτους δικαίου, που κατά τη γνώμη μου έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα προσπαθήσουμε με την Επιτροπή να προσφέρουμε μια πραγματική προστιθέμενη αξία στην έκθεση της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων. Ε, αυτή είναι η πρώτη παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης. Η διορία για τις ε, τροπολογίες λήγει 5 Μαρτίου. Θέλω να ε, συναντηθούμε δύο φορές με τους σκιώδης ηγητές για να συζητήσουμε το περιεχόμενο. Επίσης, στις 19-20 Μαρτίου θα παρουσιάσουμε τις τροπολογίες και 12 Απριλίου θα γίνει η ψηφοφορία σε εμά και 24 Απριλίου στην Επιτροπή Γιούρι. Είναι αρκετά στενό το χρονοδιάγραμμα, αλλά δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το Μάιο την, τον πίνακα αποτελεσμάτων για το 2018, καλό θα ήταν, μάλλον 17 είναι η ομιλήτρια, να προλάβουμε και εμείς προηγουμένως να διεκπαιρώσουμε το ζήτημα του πίνακα του 2017. Ε, καλώς. Περνάμε στους και ηγητές. να γενομένης από τις κυρίες Μετσόλα. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ τον κύριο Ράντεφ εδώ στη συζήτηση γιατί κολλείται σήμερα. Το θέμα του πίνακα αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντικό εργαλείο που δίνει στις επιχειρήσει και του πολίτε καλύτερη εικόνα τη αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων. Στόχο έχει την ενίσχυση τη συνεργασία και τη ανταλλαγή των πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Και θεωρούμε ότι μια αποτελεσματική, ανεξάρτητη και διαφανή δικαιοσύνη έχει θεμελιώδη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία ενό δημοκρατικού συστήματο και μια οικονομία τη αγοράς. Ε, ο σκέφτης ηγετής εκτιμά τις ε, ιστορικές διαφορές τη διάρθρωσης των συστημάτων δικαιοσύνης των κρατομέλων, αλλά θεωρούν αυτές οι διαφορές θα πρέπει να εμποδίσουν τα κρατημέλη από την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας προσφέροντα δικαστικέ αποφάσει στο κοινό, κάνοντα τι προσιτέ στο κοινό. Επίση, ο πίνακα αποτελεσμάτων αποτελεί σύστημα του Ευρωπαϊκού ε, Μηχανισμού ε, δημοκρατία, θεμελιωδών δικαιωμάτων και κράτου δικαίου, που θα δίνει μια καλή εικόνα τη κατάστασης κράτου δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη, σύμφωνα φυσικά με την αρχή τη επικουρικότητα και με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Και συμφώνουμε, στηρίζουμε από αυτήν την άποψη την έκθεση, την γνωμοδότηση. Αυτό εκ μέρου του κυρίου Ράντεφ που είναι ο σκιώδη συγγητή μα. Εκ μέρου των φιλελευθέρων τώρα η Σοφίντφελτ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ με την εισηγήτρια την κυρία Κιγιόμ για την πολύ αξιόλογη γνωμοδότησή της ε, που περιλαμβάνει πολλά εύστοχα σημεία. Θα υποβάλουμε και εμείς κάποιες προτάσεις και ενδεχομένως θα καταθέσουμε και σχετικές τροπολογίες. Ο πίνακα αποτελεσμάτων τη δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά θα πρέπει να το επεξεργαστούμε περαιτέρω, να το τελειοποιήσουμε κάπω, γιατί μέχρι στιγμή παρά είναι θεωρητικό και ακαδημαϊκό αυτό το εργαλείο. Βέβαια, ίσως επειδή τις πληροφορίες τις δίνουν τα ίδια τα κρατημέλη και τα αποτελέσματα. Και η αυτοκριτική που κάνουν τα κράτη-μέλη δεν είναι πάντα ενδελεχής. Καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τη δική της αξιολόγηση χρησιμοποιώντας και άλλες πηγές. Για παράδειγμα, την κοινωνία των πολιτών ή κάποιους ε, συνεταιρισμούς ενώσεις πολιτών που επηρεάστηκαν οι επιχειρήσεις να μην επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στις πηγές των κρατών μελών, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκέντρωση των στοιχείων για τον πίνακα αποτελεσμάτων. Επίσης, ε, είμαι ευγνώμων για ε, το ότι αναφέρατε το σύμφωνο των θεμελιωδών δικαιωμάτων δημοκρατίας και Κράτου δικαίου του Οκτωβρίου του 2016 και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για την εποπτεία σε ό,τι αφορά την πολυφωνία των ΜΜΕ. Θα ήθελα λοιπόν να προτρέψουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδέσει τις δύο εκθέσεις γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή της για έναν ευρύτερο μηχανισμό στα τέλη του έτους, αλλά του χρόνου θα μπορούσε να συνδέσει όλες αυτές τις εκθέσεις που έχουν κάποια πτυχή κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τέλος... Μια παρατηρήση που μου διαφεύγει δυστυχώς. Πάντως, είναι σημαντικό ο πίνακας αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη να διαβριθεί και να περιλαμβάνει και άλλους τομείς. Η συγκεκριά το ανέφερε σε κανένα δύο παραγράφους της γνωμοδότησής της. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ακόμη πιο σημαντικό αυτό το εργαλείο. Γιατί αν πραγματικά επισημάνει τα ε, προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και που συχνά τα συζητούμε, θα είναι ακόμη πιο σημαντικό ο πίνακα αποτελεσμάτων και θα τραβήξει και μεγαλύτερη προσοχή. Και η Τζούντιθ Σαρχεντίνη για του πράσινου. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την ε, Σιλβί Γκυγιόμ ε, για την γνωμοδότηση αυτή. Προσπάθησα λίγο να εξοικειωθώ με τα αποτελέσματα του περσινού πίνακα βαθμολογίας. Ήταν εκπαιδευτική εμπειρία. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την Σοφή και την Σιλβί ότι ίσως είναι κάπως ακαδημαϊκή υπόθεση και θα ήθελα από μια ποσοτική να περάσουμε σε μια πιο ποιοτική ανάλυση. Γνωρίζω βεβαίως ε, πως ε, ακόμα είναι εν αλλά ακριβώς ταιριάζει στο πρόβλημα. Βασιζόμαστε σε δεδομένα όχι μόνο από τα κράτη-μέλη, αλλά από ε, όργανα τα οποία δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και εργαζόμενοι στην έκθεσή μου για την Ουγγαρία παρατήρησα το ίδιο χαιρόμαστε να χρησιμοποιούμε την κρίση και ανάλυση των άλλων για να μην ε, εκφέρουμε κρίση εμείς. Α, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό γιατί γιατί σημαίνει πως ε, αν συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στην ανάλυση των άλλων ε, δεν τολμάμε να πούμε ο ένας τον άλλον την αλήθεια. Και βεβαίω παρατηρώ ότι πολλά στοιχεία για την Πολωνία εδώ πέρα λείπουν. Τώρα δεν είναι η στιγμή να αναρωτηθούμε γιατί, αλλά προξενεί εντύπωση. Θέλουμε να αντιληφθούμε την κατάσταση της δικαιοσύνης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μία χώρα που μας ανησυχεί λείπουν ε, πολλά δεδομένα. και μια χώρα η οποία φαίνεται ότι δεν έχει δεδομένα ε, είναι όπως η Κύπρος. Γιατί μάλλον δεν έχει. Ε, ενημερώθηκα, χρήσιμο, αλλά μετά ανακύπτουν άλλα ερωτήματα για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Ε, σύμφωνα λοιπόν με τη Σιλβίκη Γιώμα ότι πρέπει να εστιάσουμε στο κράτος δικαίου και τις δυνατότητες ε, να αυξηθεί και η γνώση μας ε, και ο λόγος μας επί του θέματος. Σκέφτομαι τι τροπολογίες πρέπει να υποβάλουμε. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα πάντως. Ευχαριστώ. Το Judith, αυτά που και η κυρία Κιέγγε. Ευχαριστώ Κλόντ, ευχαριστώ και εγώ την Σιλβίγκη Γκυγιόμ για την έκθεση αυτή που είναι πολύ σημαντική. Εγώ δύο πράγματα θα ήθελα να υπογραμμίσω. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο αφορά την παράγραφο που μιλάει για τον σεβασμό του κράτους δικαίου, απειλές στις θεμελιώδεις ελευθερίες κτλ. Θεωρώ ότι θα πρέπει και μέσω αυτού του εγγράφου να δούμε τι θα γίνει και με την εφαρμογή των νόμων που υπάρχουν όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων. Κατά κανόνα δεν εφαρμόζονται ποτέ και κάτι το οποίο είναι σκανδαλώδες ειδικά και στην δική μου περίπτωση όπου το έχω ζήσει πραγματικά δηλαδή στο δέρμα μου και αναγκάστηκα εγώ στο πετσί μου αναγκάστηκα ακριβώς ε, να ενημερώσω πολλές φορές ε, τους δικαστές για τους νόμους που ισχύουν ε, όσον αφορά τα ρατσιστικά εγκλήματα. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε άνοδο και πρέπει να αναπτυχθεί μια κουλτούρα για να προστατεύσουμε τα άτομα αυτά τα οποία το χρειάζονται. Το άλλο θέμα το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ακριβώς το θέμα των διαφορών που υπάρχουν όσον αφορά την απόκτηση της υπηκότητας. Ένα πρόβλημα για πάρα πολλά άτομα, για πρόσβαση σε διάφορα πράγματα θεμελιώδη, όπως η αγορά εργασίας ή μια θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα ή πρόσβαση στη στέγαση. Βλέπουμε πως υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές ε, και θα πρέπει να ενημερωθεί η δικαιοσύνη και τα δικαστήρια και σε τέτοια ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Juan Fernando. Ευχαριστώ. Θυμόμαστε όλοι ότι θεωρήσαμε όλοι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα του πίνακα ε, Βαθμολογία δικαιοσύνης. σα ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την έκθεση, είναι πολύ επίκαιρη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σκεπτικό ε, βάσει του οποίου θα, θα καταρτίζουμε αυτές τις εκθέσεις και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που με αντικειμενικό τρόπο συστηματοποιούνται σε αυτά τα έγγραφα του πίνακα για τη δικαιοσύνη. Οι επιπτώσεις των δικαστικών μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί σε μια σειρά από κράτη-μέλη ε, και που έχουν αναγνωριστεί από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και που μας έχουν οδηγήσει σε έκφραση της ανησυχίας μας αλλά και μια πολιτική αξιολόγηση από την Επιτροπή μας. Υπάρχουν κάποιες δικαστικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες πλήττουν ε, αυτή την, την αξιολόγησή μας ε, πέραν των αντικειμενικών στοιχείων που περιλαμβάνει αυτός ο πίνακας. Δεύτερο σημείο. Ναι, ορθώς επισημαίνουμε τη σημαντικότητα της ε, δικαστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θεωρώ όμως ότι θα ήταν χρήσιμο να φωτίσουμε και το είδος της εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μπορεί κανείς να γίνει ε, δικαστής. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να δώσουμε τη δέουσα σημασία σε αυτή τη διάσταση ποια θα μπορούσε να είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μιας κουλτούρας κράτους δικαίου και εκπαίδευσης όσον αφορά την εξασφάλιση και την τήρηση ευρωπαϊκών προτύπων στην δικαστική εκπαίδευση που προβλέπεται από τις εθνικές ένομες τάξεις προκειμένου να γίνει κανείς δικαστής. Γιατί υπάρχουν διαφορές συμπεριλαμβανομένων χωρών που ε, ανήκουν στην ίδια νομική οικογένεια την υπηρετική οικογένεια, για παράδειγμα Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ιταλία. Έχουμε κάποιες κοινέ αξίες και πρακτικές όσον αφορά την, ε, την, ε, τους, τους διαγωνισμούς, τις εξετάσεις που ε, υπάρχουν για να γίνει κανείς δικαστής. Αλλά στο ζήτημα της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών όσον αφορά την την, ε, την, ε, την εφαρμογή και την παροχή αυτών των αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης που απαιτούνται για να γίνει κανείς δικαστής ε, παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές και αυτό σχετίζεται και με μεγάλες κοινωνικές διαφορές όχι μόνο όσον αφορά το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο των ανθρώπων που επιδιώκουν να γίνουν δικαστές αλλά και από άποψη φίλου για παράδειγμα. Θέλω λοιπόν να πω ότι ε, θα ήταν ε, καλό και θα άξιζε τον κόπο και αυτές οι διαστάσεις να συμπεριλαμβάνονται στην τελική μας έκθεση. Τόμας. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Εδώ, εδώ πίσω είμαι. Ίσως δεν με είχατε δει νωρίτερα. Προσωπικά έχω διάφορα σχόλια που θα ήθελα να κάνω για αυτή την έκθεση. Πρώτον, κάτι που ανέφεραν και άλλοι τα στοιχεία με τα οποία τροφοδοτείται αυτός ο πίνακας. Η έκθεση αυτή είναι άχρηστη. Θα μπορούσα να την είχα συντάξει εγώ μέσα σε 10 λεπτά. Θα μπορούσα να είχα ε, αναζητήσει τα αρχικά δεδομένα ε, online. Όλα αυτά είναι γνωστά. Αν μάλιστα ε, έχετε απλά αντιγράψει την έκθεση αυτή από τις προηγούμενες χρονιές και αλλάζατε την εφερμηνία, ε, δεν θα υπήρχε καμία διαφορά. Τα έχουμε ε, επικρίνει αυτά τα στοιχεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλουμε θεωρητική έκθεση η οποία δεν θα προσθέτει τίποτα. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι θέλουμε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των, των στοιχείων. Και βλέπω εδώ όλες αυτές οι γραφικές αναπαραστάσεις. Τι συγκρίνουν εν τέλει. Ε, δείτε τις εξηγήσει που, δίνονται. Μας, μας αγνοούν ε, ως προς τις ε, επικρίσεις που έχουμε κάνει και τα στοιχεία, τα σχόλια που έχουμε υποβάλει. Θέλουμε να πούμε στην Κομισιόν ότι δεν θέλουμε να λαμβάνουμε τέτοιες άχρηστες εκθέσεις. Δεν, ε, δεν έχουν καμία αξία τέτοιου είδους εκθέσεις στην εποχή της ψηφιοποίησης και του διαδικτύου. Προφανώς κάποια κράτη-μέλη δεν υποβάλλουν όλα τα στοιχεία που έχουμε. Σε κάποια κράτη-μέλη δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά στοιχεία. Σε κάποιες, κάποια άλλα κράτη-μέλη όμως υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων. Πού υπάρχει σύγκριση, πού είναι τα δεδομένα σε αυτή την έκθεση. Ε, ε, εγώ βλέπω σε αυτή την έκθεση ε, εντυπώσεις και μόνο, εκτιμήσεις, καθόλου στοιχεία. Μπορώ να διατρέξω τα, τις σελίδες μία προς μία είναι γελίο. Για παράδειγμα, ε, το, το, το κομμάτι που αφορά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών. Δεν υπάρχει καν, δεν, δεν υπάρχει πληροφορία, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την εκπαίδευση που λαμβάνουν οι δικαστές προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Αλλά και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Συνήθως ε, οι δικαστές μπορεί να παραμείνουν στη θέση τους για 30 χρόνια και στη διάρκεια αυτών των 30 ετών μπορούν να λαμβάνουν εβδομάδες εκπαιδεύσεων. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στην έκθεση. Νομίζω ότι είναι πραγματικά γελία αυτή η έκθεση, γελάω δηλαδή. Ε, συγκρίνουμε πράγματα ασύγκριτα και νομίζω ότι η έκθεση με τον τρόπο που έχει ε, συνταχθεί είναι άχρηστη, δεν έχει νόημα κανένα. Είναι πραγματικά... Ε, ε, γεγονός ότι δεν χρειάζεται, κανείς δεν χρειάζεται τέτοιου είδους εκθέσεις. Ε, κύριε Τόμας, έχετε κακό πρωινό μάλλον, έχετε κακή διάθεση σήμερα. Όχι. Ναι, όχι, ναι. Αλήθεια, γιατί και την περισμένη φορά είχα εξοργιστεί με τη συζήτηση. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτή η επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, ε, Σημειώνουμε πάντω τι επικρίσεις. Δεν ξέρω, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να παρέμβει πριν ε, επανέλθουμε στην εισηγητριά μα την κυρία Σιλβί Γιώμ. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Έχω σοκαριστεί από την τελευταία παρέμβαση. Όταν ένα ευρωβουλευτή δηλώνει ότι ο πίνακα αποτελεσμάτων του, του προκαλεί γέλο τάπ, πραγματικά ε, μα σοκάρει. Γιατί φάνηκε από τη συζήτηση ότι είναι χρήσιμο εργαλείο ο πίνακα αποτελεσμάτων και μάλιστα έχει στόχο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δικαστικών του συστημάτων. Και γνωρίζουμε όλοι ότι μια αποτελεσματική δικαιοσύνη έχει κέρια σημασία για το σεβασμό του κράτους δικαίου και γι' αυτό θεωρούμε ότι ο πίνακα αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στο σεβασμό του κράτου δικαίου και στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία που δεν προέρχονται μόνο από τα κράτη-μέλη. Χρησιμοποιούμε στοιχεία και από τα δίκτυα δικαστών, από διαφορετικές επιτροπές και γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να γεφυρωθεί το κενό που έχουμε στη συλλογή δεδομένων, αλλά κάθε χρόνο σημειώνουμε πρόοδο και συγκεντρώνουμε όλο και περισσότερα στοιχεία. Είναι αλήθεια ότι κάποιες χώρες τις προηγούμενες χρονιές έδιναν λιγότερα πιο φιδωλά τα στοιχεία, αλλά για το 2018, για τον πίνακα αποτελεσμάτων του 2018, που θα δημοσιευθεί ως ο στα μέση της Άνοιξης τέλος πάντων, θα δείτε ε, και νέα στοιχεία από την Πολωνία. Οπότε υπάρχουν στοιχεία και για τη χρήση των μέσων ε, και των, πληροφοριών, των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας και ως τέτοια είναι αξιόπιστα. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ε, τα καταγράψαμε πισταμένος και περιμένουμε και την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που είναι αρμόδια κατ' ουσία. Νομίζω ότι είναι επικοδομητική η κριτική του πίνακα αποτελεσμάτων από τα μέλη της Επιτροπής και αυτό το νόημα έχει και η συζήτηση και όλα θα τα λάβει υπόψη αυτά η συγγήτρια. Και μπορεί να μην είναι τέλειος ο πίνακας αποτελεσμάτων, αλλά όσα είναι είναι πολύ σημαντική. Η κυρία Ιντβελτ. Εγώ διαφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι ότι υπάρχει κενό ε, στη συλλογή των πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει να αποκλείσει κάποιε πηγέ. Είναι πολιτική επιλογή από ποιε πηγέ συγκεντρώνει τι πληροφορίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μπορεί να λέμε ότι το διπλωματικό ή γραφειοκρατικό καθεστώς της ε, παρελθόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κατανοητό. Αλλά είμαστε σε μια πολιτική ένωση ε, θα πρέπει να κάνετε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των εθνικών δικαστικών συστημάτων και να μην επαφίεστε μόνο στις πληροφορίες των εθνικών αρχών. Φυσικά θα ρωτήσετε και τις εθνικές αρχές, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και άλλες πηγές από άλλους φορείς. Και είναι η πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από ποιες πηγές θα συλλέξει τις πληροφορίες της. Όπως είπα, κάποιοι σκιώδεις ε, εισηγητές σχολίασαν και τις άλλες πηγές. Ε, αναφερθήκατε στο Σύμβουλο της Ευρώπης. Οπότε η συγγήτρια τα σημειώνει όλα αυτά. Θα τα λάβει υπόψη. Βέβαια, ο χρόνο είναι ελάχιστο. Μόνο δύο συνεδριάσει και οδόνηση για τον θα γίνουν. Δεν ξέρω, Σιλβί, κάνε μια προσπάθεια να ανακεφαλαιώσει και να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, θα μπορούσαμε να είχαμε ε, κοιμηθεί, αλλά όχι. Τελικά ήταν πολύ πιο ζωηρή συζήτηση από ό,τι ε, αναμέναμε. Πολύ ενδιαφέρον συζήτηση μεταξύ πολιτικής και γραφειοκρατίας και μερικές φορές η υποκειμενικότητα ή η αντικειμενικοτητα ε, που χαρακτηρίζει τις εκθέσεις, όπως είπε ο Τόμας. Υπάρχουν και κάποια μέσα που δεν αφορούν την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα. Όντως, ε, ε, αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, περιλαμβάνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων, Τόμα. Δεν ήταν σωστό αυτό το σχόλιο. Ε, είπατε ότι ήταν κάπως στήρο αυτό το έγγραφο. Δεν είναι ε, όντως πολύ πρακτικό, είναι κάπως ακαδημαϊκό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και άγωνο, ότι είναι στήρο, γιατί δεν είναι αρκετά σαφή εικόνα για τα διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία. Ε, έγιναν αρκετά εύλογα σχόλια και πολύ θεμητά από τους συναδέλφους και ε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο το κράτος δικαίου, όπως είπα και εγώ αρχικά στην παρέμβασή μου. Επίσης, ε, σημείωσατε ενδιαφέροντα σχόλιά σας για τον τρόπο ανάπτυξης των δεδομένων και τις προτάσεις που θα κάνουμε στα κράτη-μέλη ή πώς μπορούν να επηρεάσουν τα δικαστικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Για να μην μακρηγορήσω και παρατείνουμε τη συζήτηση, μην ξεχνάτε ότι η γνωμοδότηση είναι πολύ σύντομη εκφύσεως, οπότε περιμένουμε τις τροπολογίες για να την επιμηκύνουμε κάπως και για να την καταστήσουμε πιο στιβαρή και πιο αυστηρή. Ε, θα κάνω και εγώ κάποια σχόλια για την ποινική δικαιοσύνη. Αυτή είναι στιγμή με τις τροπολογίες σας να εμπλουτίσετε τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Okay, we're in very good hands with our part of the... Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι. 5 Μαρτίου είναι η προθεσμία της τροπολογίας. Ε, πολύ συγγνώμη. Σας ευχαριστώ όμως ε, και πάλι για τις ε, παρεμβάσεις σας στην συζήτηση, παρεμβάσεις με πάθος. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 16, το οποίο αφορά την Ελβετική Συνομοσπονδία και το σχετικό δημοψήφισμα για την ελεύθερη κυκλοφορία. Με χαρά καλωσορίζω τον πρέσβη τον κύριο Μπούχερ. Α, έρχεται.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 Okay, colleagues, we come to point 16. Uh, λοιπόν, περνάμε στο σημείο 16, το οποίο αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Χαίρομαι που έχει έρθει μαζί μας ο κύριος Μπούχερ, επικεφαλής Ελβετικής Αποστολής στην Ένωση. Ζήτησαν οι συντονιστές ε, την ενημέρωση για το τι έγινε μετά το ελβετικό δημοψήφισμα. Αν αναρωτιέστε γιατί μας απασχολεί λοιπόν το θέμα το δημοψήφισμα, όπως ε, θα θυμούνται οι συνάδελφοι, έγινε στις 9 Φεβρουαρίου και θα θυμάστε ότι η πλειοψηφία του ελβετικού λαού ζήτησε να εισαχθεί ένα σύστημα ποσοστώσεων ε, για επικόους άλλων χωρών. Ξέρουμε ότι αυτό βεβαίως ε, δεν συμβιβάζεται με το καστός της ελεύθερης κυκλοφορίας για τις χώρες που μετέχουν στην ενιαία αγορά. Τώρα θα ακούσουμε λοιπόν μια σύντομη δήλωση από τον κύριο Πρέσβη που θα μας ενημερώσει πώς ε, προχωράει η κατάσταση και ποιες είναι οι πιθανές ε, λύσεις. Μετά θα γίνει μια σύντομη συζήτηση με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επίσης και την Κομισιόν. Κύριε Μπούκερ, Μπούχερ, έχετε τον ε, λόγο. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, ε, κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μα δίνετε αυτό το βήμα για συζήτηση σήμερα. Για να καθορίσω το πλαίσιο, επιτρέψατε μου να αναφέρω το πρόφανες. Η Ελβετία έχει πολύ στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεωγραφικούς, ε, πολιτισμικούς και οικονομικούς Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο σημαντικότερος μακράν ε, εμπορικός εταίρος μας ε, και η Ελβετία είναι ένας εκ των τριών σημαντικότερων εταίρων της Ένωσης ε, μετά της ΙΠΑ ε, και την Κίνα. Έχουμε μια σειρά συμφωνιών αυτή τη στιγμή. Είμαστε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας που αντιμετωπίζει τα θεσμικά ζητήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ε, πρόσβασης ε, στην αγορά. Η Ελβετία παραμένει προσιλωμένη σε αυτή τη διαδικασία με μια λύση η οποία θα σέβεται την κυριαρχία της Ελβετίας λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαιότητες ε, της εσωτερική αγοράς προς το συμφέρον και της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελεύθερη κυκλοφορία που είναι το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης είναι άλλο ένα παράδειγμα των στενών δεσμών που έχουμε πάνω από 464.000 Ελβετοί πολίτες κατοικούν σε χώρες ΕΟΚ και ΕΖΕΣ και στην Ελβετία έχουμε πάνω από 1,4 εκατομμύρια πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΖΕΣ. Επιπλέον πάνω από 300.000 άτομα διασχίζουν τα σύνορα κάθε μέρα για να εργαστούν. Όμως, εάν η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ευκαιρία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει και προκλήσεις, όπως ε, ο αυξημένος ανταγωνισμός αγοράς εργασίας, ειδικά σε μεθοριακές περιοχές, η φόβια θέμη του ανταγωνισμού και του να μείνουν εκτός ε, οι ε, γηγενείς και βεβαίως η ανάγκη διατήρησης των κοινωνικών προδιαγραφών και προδιαγραφών απασχόλησης. Ο ελβετικός λαός εξέφρασε τις ανησυχίες τους στο σχετικό δημοψήφισμα, ανησυχίες που υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως δείξε η τελευταία συζήτηση. Βεβαίω ε, τα θετικά αποτελέσματα είναι ένα προαπαιτούμενο για μια ανοιχτή κοινωνία και για την αποδοχή της ελεύθερης κυκλοφορίας. Τώρα θα ήθελα να σας εξηγήσω την εφαρμογή της Πρωτοβουλία τη 9 Φεβρουαρίου κατά της μαζικής μετανάστευση όπως λέγεται. Στις 9 Φεβρουαρίου 2014 η πρωτοβουλία εγκρίθηκε από το 50,3% των ψηφοφόρων στα περισσότερα καντόνια για να εφαρμοστεί η νέα συνταγματική διάταξη, το άρθρο 121α του Ελβετικού Συντάγματος εγκρίθηκε από την Βουλή αναθεώρηση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών που συμφωνεί πλήρως με την ελεύθερη κυκλοφορία. Οι λεπτομέρειες ε, κατόπιν εγκρίθηκαν ένα έτος αργότερα από την κυβέρνηση, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, το Δεκέμβριο του 2017 και ο αναθεωρημένος νόμος θα τεθεί ισχύ την 1η Ιουλίου φέτος. Να τονίσω ότι μέσω της ε, διαδικασίας αυτής ε, και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η Ελβετία σεβάστηκε τις υποχρεώσεις της ε, και λειτουργούσε ανα πάση στιγμή η Συμφωνία περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Οπότε σεβόμασταν τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Οι αριθμοί ε, δείχνουν το πόσο καλά λειτουργεί η Συμφωνία περί ελεύθερης κυκλοφορίας ε, προσώπων. Από όταν ετέθη ενισχύ το 2002 η μετανάστευση από τις ευρωπαϊκές χώρες προς την Ελβετία αυξήθηκε κατά πολύ. Όπως ανέφερα, αυτή τη στιγμή 1,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν στην Ελβετία και αυτό είναι το 17% του πληθυσμού της χώρας. Ο πληθυσμός της Ελβετίας αυξήθηκε στο διάστημα αυτό από 7,3 σε 8,4 εκατομμύρια. Αυτό είναι ε, ε, το 1 το ένα δέκατο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του χώρου ΕΖΕΣ που εργάζονται σε άλλη χώρα. Δηλαδή η Σουηδία με τα 8,4 εκατομμύρια κατοίκους αντιπροσωπεύει το 10% της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. Και ο αριθμός επίσης ε, των ε, μεθοριακών ε, εργαζομένων διπλασιάστηκε από τα ετέθη ενισχύ συμφωνία και όπως σας είπα τώρα φτάνει τα 300.000 άτομα. Τι έχει γίνει. Η νομοθετική πρωτοβουλία περιέχει στοχευμένα μέτρα κατά της ε, ανεργίας ε, και ενισχύει την απασχόληση στην Ελβετία περιλαμβανομένων των πολιτών της Ένωσης. Συγκεκριμένα ο θεωρημένος νόμος εισάγει μία υποχρέωση να κοινοποιούνται στα τοπικά γραφεία εργασίας ή ε, προσφορές εργασίας όταν φτάσουμε ένα όριο ανεργίας, αυτό το οποίο θα είναι 8% από τον Ιούλιο και 5% από 1η Πρώτου 2020. Επιπλέον, όσοι ε, είναι άνεργοι θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, 5 εργάσιμες ημέρες και κατόπιν μπορεί να δημοσιευθεί η αγγελία πέραν των τοπικών γραφείων εργασίας. Όλα τα άτομα τα οποία έχουν εγγραφεί σε ένα τοπικό γραφείο εργασίας, ανεξαρτήτως υπηκότητας, μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο. Αυτό περιλαμβάνει τους ε, υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΖΕΣ που κατοικούν στην Ελβετία ή αναζητούν εργασία στην Ελβετία. Η απέτηση κοινοποίησης όπως ε, και η πρόσβαση των ε, ανέργων σε αυτές τις ε, πληροφορίες θεωρούμε ότι είναι ένα δικαιολογημένο μέτρο για να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Συνοψίζοντας, η εφαρμογή της συνταγματικής διάταξης έχει απασχολήσει εδώ, απασχολεί εδώ και τρία χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία. Η Ελβετία, όπως ξέρετε, είναι πολύ υπερήφανη για την άμεση δημοκρατία που επιτρέπει στους πολίτες να εκφράσουν τις ανησυχίες της και η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο μετά βρίσκουν συμβαστικέ λύσεις που βρίσκονται ακριβώς στην βάση του ελβετικού κοινωνικού συμβολέου, της σταθερότητας και της ευημερία. Με την πρωτοβουλία αυτή καταφέραμε να βρούμε μια λύση η οποία σέβεται πλήρως ε, την Συμφωνία Ελεύθερης Κυκλοφορίας και αντιμετωπίζει τις θεμητές ανησυχίες ε, των εργαζομένων όχι μόνο στην Ελβετία αλλά ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η λύση είναι η μη διακριτική μεταχείριση, καθώς οποιοδήποτε αναζητεί εργασία στην Ελβετία μπορεί να εγγραφεί σε ένα γραφείο εργασίας. Δεν γίνεται διάκριση με βάση την υπηκότητα και άρα δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Δεδομένου του ότι αυτή η διαδικασία πλέον ολοκληρώθηκε, αναμένουμε την συνέχεια του ανοιχτού και επικοδομητικού διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Ωραία. Έχουμε μέχρι τις 11 και 4 χρόνο για το θέμα αυτό, οπότε ε, θέλω να ρωτήσω την ομίγυρη ποιος θέλει το λόγο. Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον γιατί το ζήτησαν οι συντονιστές να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι Μπεν Νοκνό από την ΕΕΘ και έχουμε από τη Γενική Διεύθυνση για τη Δικαιοσύνη και την Απασχόληση εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια σύντομη επισκόπηση της αξιολόγησης της κατάστασης να υπενθυμίσω ότι στη Συμφωνία για την Ελεύθερη Διακίνηση Προσώπων, η Ελβετία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν για την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, ε, συμπεριλαμβανομένη τη εισόδου, διαμονή, πρόσβαση σε εργασία, άσκηση ανεξάρτητων δραστηριοτήτων και προοχή υπηρεσιών με ίσους όρους όπως και οι Ελβετοί πολίτες. Επίσης προβλέπεται συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών σπουδών και προσόντων στις αιτήσει ε, συναδρία της Κοινής Επιτροπής για τη διαχείριση της συμφωνίας έχουμε ε, αποπτεύσει και ε, εξετάσει τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και μετά την υιοθέτηση του νόμου περί του 2016 και την τροποποίηση που έγινε που ανέφερε ο πρέσβη. είχαμε έκτακτη συνεδρία Συμμεκτής Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2016 για να διευκρινίσουμε κάποιε πτυχέ αυτής τη νομοθεσία. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του περιορισμού που επιβάλλει στην πρόσβαση των πληροφοριών για τι ε, θέσει απασχόληση και τον ορισμό των κριτηρίων για τα κατόφλια και του ε, τομεί, ε, επαγγελματικέ ομάδε ή τι περιφέρειες στι οποίε ισχύουν αυτά τα κατόφλια εκφράσαμε τις ανησυχίες μας κυρίως για τους όρους και τις δυνατότητες των Ευρωπαίων πολιτών να καταγραφούν σε ευρωπαϊκά, ε, σε ευρωπαϊκά γραφεία εργασία. Ενώ η Ελβετία μας διαβεβαίωσαν ότι υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητα από τη διαμονή η προηγούμενη απασχόληση για τους Ευρωπαίους πολίτες. Οπότε και οι αναζητούντες απασχόληση, οι Ευρωπαίοι πολίτες που μετέβησαν στην Ελβετία και που ψάχνουν δουλειά μπορούν να καταγραφούν στα γραφεία εργασίας της Ελβετίας. Επίσης, ε, τα πρόσθετα μέτρα που μπορούν να υποβάλουν τα, κατώ, καντόνια ε, που δεν, είναι, δεν μπορούν να παραβιάζουν τη Συμφωνία για την Ελεύθερη Διακίνηση των Προσώπων. Και από τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου του 2017, το σχέδιο πρότασης ε, εξετάστηκε στην ε, Μικτή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2017. Και πάλι διευκρινίσαμε κάποια θέματα και παρουσιάσαμε τις ανησυχίες μας ότι αφορά το στόχο των κυρώσεων που προβλέπονται, τη μέγιστη διάρκεια ε, ισχύω των περιορισμών στην πρόσβαση των πληροφοριών και άλλες πιθανές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες, όπως ε, υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και δικαιολόγησης. Πάντως οι απαντήσεις Ελβετίας ήταν καθυσχαστικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τα αποτελέσματα της Επιτροπής και της ΕΕΤ είναι τα εξή. Με βάση το γράμμα του κειμένου και της των εφαρμοστικών διατάξεων θεωρούμε ότι ο νόμος αυτός μπορεί να επηρεαστεί χωρίς να παραβιάζονται τις υποχρεώσεις της Ελβετίας ό,τι αφορά τη Συμφωνία της Ελεύθερης Διακίνησης των Προσώπων. Βέβαια, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες όπως ξέρουμε. Οπότε θα συνεχίσουμε την στενή παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών και από τα τοπικά γραφεία και από από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή ο νόμο τον Ιούλιο του 2018, ώστε να αποφευθούν διακριτική μεταχείριση βάρο των Ευρωπαίων πολιτών ή παραβίαση του δικαιώματός του για ελεύθερη διακίνηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία τη Δράσης για την παρέμβασή τη. Κυρία Μετσόλα, ε, μιας και οι συντονιστές ζήτησαν να υπάρξει συζήτηση για αυτό το θέμα θα ήταν καλό να παρέμβουν κιόλα. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρέσβη για την παρουσία του εδώ και την ενημέρωσή του σχετικά με ορισμένες ανησυχίες που έχουμε εκφράσει ως προς την ερμηνεία κάποιων νομικών, νομοσχεδίων και νομικών πράξεων που έχουν ε, υποβληθεί τα τελευταία χρόνια. Για μας η ελεύθερη κυκλοφορία είναι αδιαπραγμάτευτη και όπως είπε και ο εκπρόσωπος ΕΙΕΔ υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν και που έδωσαν την εικόνα ότι δεν ήταν η βασική αρχή ε, η ελεύθερη κυκλοφορία που ε, τα διέτρεχε, ε, ιδίως όσον αφορά την αναζήτηση εργασία, τα άτομα που αναζητούν εργασία, υπήρχαν ανησυχίες δια, διακριτική μεταχείριση εις βάρος ε, Ευρωπαίων πολιτών ή εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο ε, λιγότερο διαφανή σε σύγκριση με τους Ελβετούς πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, απεκατέστησες ε, την αξιοπρέπεια του σώματος των συντονιστών. Είναι, είναι ένα από αυτά τα ζητήματα που ήταν πολύ καυτά και ε, Μια και η δική μα Επιτροπή επιφορτίζεται με το να επεξεργαστεί ε, το 40% των νομοθετικών προτάσεων της θητείας αυτής, ε, ήταν πραγματικά καιρός να γίνει αυτή η συζήτηση. Είναι δύσκολο βεβαίως να υπάρχει πάντοτε σήμερα ειδικά ήταν δύσκολη η φυσική παρουσία των συντονιστών. Βεβαίως θα καταγράψαμε όλα αυτά τα στοιχεία που μας είπατε. Είναι ε, είναι πηγή ανησυχία. Νομίζω ότι κύριε Πρέσβη απαντήσατε σε πολλά από τα θέματα. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για την παρουσία της και την ε, κυρία Μέτσολα. Αν θέλετε να απαντήσετε στο, στο ερώτημά τη και να παρέμβετε ή να τοποθετηθείτε για οτιδήποτε άλλο που ίσως δεν καλύψατε ε, εισηγητικά, έχετε το χρόνο να το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η κίνηση αυτή είναι άλλη μια συμβολή στην εξομάλυνση των σχέσεών μας, όπως είπα και το εισηγητικά, οι δεσμοί Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικοί και υπάρχει και περιθώριο ανάπτυξης των δεσμών αυτών. Πρέπει να καταβάλουμε και οι δύο πλευρές κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ ε, για την παρουσία σας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επίσης. Ευχαριστούμε συνάδελφοι και θα παρακολουθούμε βεβαίως ε, το ζήτημα αυτό στενά και θα ενημερώσω για τα, τους συντονιστές για όσα μας είπατε. Okay, So, colleagues, the next... Λοιπόν, συνάδελφοι, το επόμενο θέμα είναι κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γενικών και Ισότητας των Φύλων. Θα γίνει στις 11 και 4. Θα κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα έως εκείνη την ώρα, έως στις 11 και 4. Επανερχόμαστε λοιπόν 11 και 4 για να δούμε για να δούμε το θέμα της καταπολέμησης